we don't want to lose time. We start with uh, point 8 of the agenda, which is volunteering Χάσουμε χρόνο. Να έρθουμε τώρα στις ε, δραστηριότητες ε, στην Ευρώπη. Ο Μάρκος Κόρια είναι ο εισηγητής μας. Και έτσι θα του δώσω αμέσως τον λόγο. Παρακαλώ, Μάρκος. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. η έκθεση που έχω υποβάλει, που έχω εκπονήσει και μάλιστα θέλω να ευχαριστήσω εδώ την Γραμματεία για την ε, πολύτιμη βοήθειά του. Στην έκθεση λοιπόν αυτή έλεγα ότι έχω προσπαθήσει να εισάγω κάποια στοιχεία τα οποία συζητήσαμε την προηγούμενη φορά, δηλαδή στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων που είχαμε για το θέμα αυτό. Βλέπετε την έκθεσή, σας, ε, την έκθεση αυτή στο φάκελό σας. Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω όλα γιατί φαντάζομαι ότι έχετε ήδη διαβάσει την έκθεση και τώρα απλώς ε, θα πρέπει να γίνουν κάποιες επιπλέον παρατηρήσεις επ' αυτής. Θα ήθελα απλώς ε, να υπογραμμίσω κάποια στοιχεία. Την προηγούμενη φορά λοιπόν είχαμε καθορίσει έναν τρόπο λειτουργίας ε, ως εξής, ε, δηλαδή πέρα από τα σημεία τα οποία ε, επισημαίνουμε στα, για τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού να προβλέψουμε μία σειρά από σημεία και από πρωτοβουλίες έτσι ώστε ο εθελοντισμός να μην σταματήσει ή να μην σταματήσει να γίνεται συζήτηση για τον εθελοντισμό μετά το πέρας του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού ε, και ότι το ζήτημα αυτό το τόσο σημαντικό να συνεχίσει να μας απασχολεί. Συνέβησαν πολλά ενδιαφέροντα κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους ε, και έχουμε και πολλά αιτήματα τα οποία προέρχονται από ε, ομάδες εθελοντών, ενώσεις εθελοντών που ζητούν μεγαλύτερη εμπλοκή της Ευρώπης στο θέμα αυτό. Επομένως, μεταξύ των γραφωμένων μου υπάρχει και το εξής, πρόβλεψη ε, του καθεστώτος, του καταστατικού συγγνώμη, ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθελοντισμού, έτσι ώστε να έχουν μια υπόσταση και απέναντι στις ενωσιακές, στους ενωσιακούς θεσμούς και όργανα, αλλά και απέναντι στα εθνικά όργανα. Και επίσης να πούμε ότι μέσω του εθελοντισμού οι νέοι να μπορούν να μαζεύουν σημεία τα οποία θα προστίθενται στο Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων. Ε, επίσης αναφέρουμε την ανάγκη δημιουργίας του Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής ε, Βοήθειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, πρέπει να είμαστε σε θέση να δίνουμε απάντηση και στις διάφορες ανθρωπιστικές κρίσεις οι οποίες δυστυχώς έχουν αρχίσει και υπάρχουν ακόμα και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται και εσωτερικό πρόβλημα πλέον και επομένως θα πρέπει να υπάρχουν ε, και διάφορες οργανώσεις για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό. Ζητώ επίσης από τα κράτη-μέλη και από την Κομισιόν να προβλέψουν ένα ενιαίο σημείο επαφής ως ε, ε, διαρκή, διαρκές σημείο επαφής μεταξύ των οργανώσεων και των θεσμικών οργάνων. Υπογραμμίζουμε επίσης την ανάγκη δημιουργίας ε, μιας ευρωπαϊκής θηρίδας έτσι ώστε να διευρυνθούν οι γνώσεις μας ε, ε, όσον αφορά τις εθελοντικές δράσεις σε ενωσιακό επίπεδο που θα συμπεριλαμβάνει και μία τράπεζα δεδομένων των βελτίστων πρακτικών στα πλαίσια του εθελοντισμού έτσι ώστε ε, να δημιουργηθεί αλλά και να ενισχυθεί περαιτέρω αυτό το κύμα, του, το ρεύμα του εθελοντισμού. Δηλαδή να υπάρξουν οι καλές πρακτικές αλλά και αυτές οι ζυμώσεις οι οποίες θα γνωστοποιήσουν καλύτερα τα όσα γίνονται. Ε, βεβαίως, ζητούμε να διατηρηθεί ε, και ε, ο οργανισμός, το συντονιστικό όργανο το οποίο δημιουργήθηκε στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού έτους ε, και που βοηθάει και τη δράση των διαφόρων οργανώσεων επιτόπου αλλά και τον συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπογραμμίζουμε την ανάγκη οι εθνικές και περιφερειακές αρχές, οι τοπικές αρχές να απλουστεύσουν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και να δημιουργήσουν ε, ε, φορολογικά κίνητρα για τις ε, ενώσεις και επίσης εντάξαμε και την ανάγκη ασφαλιστικής κάλυψης των ε, εθελοντών που πρέπει να είναι υποχρεωτική. Το είχαμε αναφέρει και την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, ασφαλιστική κάλυψη, υγειονομική κάλυψη ε, να είναι υποχρεωτική για τις δραστηριότητες των εθελοντών και επίσης μέσω των κρατών μελών να ε, δοθεί ιδιαίτερη ε, σημασία στην ε, άτυπη αλλά και επίσημη εκπαίδευση, κατάρτιση των εθελοντών έτσι ώστε και αυτοί να είναι όσο γίνεται πιο σωστοί και υπεύθυνοι στις ε, καθημερινές τους δραστηριότητες. Αυτά σε γενικές γραμμές είναι τα κυριότερα σημεία τα οποία ήθελα να υπογραμμίσω. Υπάρχουν και άλλα, αλλά όπως είπα και εξ αρχής προτιμώ να μην ε, μακρηγορήσω αναφερόμενο σε πράγματα τα οποία ο καθένας μπορεί να διαβάσει στο φάκελο. Νομίζω ότι πέρα από την ε, ανάλυση του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί περαιτέρω και στο μέλλον να αναπτυχθεί ο τομέας αυτός. Ε, πρέπει να πούμε ότι αυτό το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού ήταν καλό, έδωσε καλά αποτελέσματα και να συνεχίσουμε στην ίδια τροχιά. Ε, περιμένω βεβαίως ε, και τις παρατηρήσεις των συναδέλφων, θα έχουμε και τις τροπολογίες, θα συζητήσουμε τα θέματα αυτά και με τους κοιόδης εισηγητές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε με όσο γίνεται πιο ενωτικό τρόπο στην ψηφοφορία. Ε, είναι ένα από τα θέματα στα οποία θα πρέπει να υπάρχει συνένεση, να εμφανιστούμε ενωμένοι και όχι μοιρασμένοι, γιατί ε, πρέπει να δώσουμε και ένα καλό θετικό μήνυμα προς όλους αυτούς τους νέους που κάθε μέρα μέσω του εθελοντισμού προσπαθούν να βοηθήσουν την κοινωνία. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Νεδαλόβα. Ε, ναι, Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον Μάρκο για την υψηλή ποιότητα έκθεσή του. Φαίνεται καθαρά ότι στο πρόσωπο του Μάρκο έχουμε έναν αληθινό εμπειρογνώμονα περί Είναι λοιπόν σημαντικό να γνωρίζουμε προς τα που κατευθυνόμαστε. Είναι μια δραστηριότητα εθελοντισμός που πρέπει να αναγνωριστεί. Ένα πέμπτο του ευρωπαϊκού πληθυσμού αφιερώνει μέρος του χρόνου τους τις εθελοντικές δραστηριότητες. Χρειάζονται προστασία. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε ορισμένα θέματα τώρα μετά από το έτος του εθελοντισμού με τη δημιουργία της συμμαχίας των εθελοντών και έχουμε, να έχουμε επιτέλους ένα όργανο το οποίο να συμβάλλει στην ανάπτυξη του εθελοντισμού στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στην χώρα μου είναι πολύ καλύτερη και μεγαλύτερη η συνειδητοποίηση για τον εθελοντισμό. Έχουμε ιστοσελίδες, όπως είπατε και εσείς, στη Σλοβακία για παράδειγμα έχουμε μία ιστοσελίδα που ε, επιγράφεται volunteering.sk. Εκεί παρακολουθεί κανείς τις ε, διάφορες δραστηριότητές τους και ανοίγονται και δυνατότητες να συμμετάσχει κανείς. Όποιος επιθυμεί μπορεί να συμβουλευτεί την ιστοσελίδα μπορεί να δει ε, ποιε οργανώσεις προσφέρουν ε, δυνατότητες ε, να συμμετάσχει σε εθελοντικές δραστηριότητες κλπ. Προ δύο εβδομάδων περίπου εγώ συναντήθηκα με εκπροσώπους εργοδοτών μεγάλων επιχειρήσεων στη Σλοβακία και αυτοί έχουν τη διάθεση να συμβάλλουν στην υποστήριξη του εθελοντισμού. Ο εθελοντισμός λοιπόν είναι σημαντικός γιατί έχει και σημασία να αναγνωριστούν οι δεξιότητες που αποκτούν οι εθελοντές κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους. Για παράδειγμα και η δραστηριοποίηση σε οργανώσεις νέων, νεολαίας κλπ. είναι και αυτές ε, τέτοιου χαρακτήρα που επιτρέπουν την ε, ε, συγκέντρωση προσόντων και ούτω καθεξής που μετά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλους τομείς. Αυτό θα ήθελα να τονιστεί λίγο περισσότερο στην έκθεση. Το άλλο που είναι σημαντικό για τον εθελοντισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το είχα πει και την προηγούμενη φορά, είναι η προστασία της υγείας, η κοινωνική προστασία και η προστασία της υγείας των εθελοντών. Να ε, φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο έστω και αν δεν τους προσφέρει πλήρη κάλυψη, να τους προσφέρει κάποια κάλυψη. Αν δηλαδή κάτι πάθουν στη διάρκεια της άσκησης των εθελοντικών τους ε, δραστηριοτήτων, να μην είναι εντελώς ακάλυπτοι πρέπει να δούμε και από αυτή την άποψη τα κείμενά μας για τον εθελοντισμό. Διότι οι χώρες μέλη φορολογούν και τις επιστροφές εξόδων των εθελοντών ή ε, αποζημιώσεις κλπ. που λαμβάνουν. Πρέπει επίσης να διατεθούν περισσότερα κονδύλια για την ανάπτυξη του εθελοντισμού στο νέο πρόγραμμα Έρασμος ΣΥΝ και προς τα εκεί θα κατευθυνθούμε με την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Προσφορά Υπηρεσιών υπέρ των νέων και για την Ευρωπαϊκή ε, Ιθαγένεια το ίδιο. Εγώ θα μπορούσα να συνεχίσω ε, θεωρητικό σε επάπειρο ε, με αυτά, αλλά δεν θέλω. Θα κάνω κάποιες τροπολογίες, αλλά θα είναι ίσονο σημασία γιατί με ικανοποιεί η έκθεση. Η Μαρή Τερέζα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μάρκο, νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να σε ευχαριστήσουμε για την ενεργητικότητα με την οποία ασχολήθηκες με αυτό το θέμα του εθελοντισμού. Ε, πρόκειται για πραγματικά μια εμπειρία πολύ θετική που ε, εμπλουτίζει και εμάς αλλά και τους νέους που βρίσκονται ενδεχομένως και σε ένα μεταβατικό στάδιο προς την απασχόληση. Ε, μέσω του εθελοντισμού μπορεί κανείς να αποκτήσει σε ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο ε, εμπειρία εργασίας. Μπορεί να βοηθήσει την ένταξη στην κοινωνική και επαγγελματική ε, ζωή. Κατά αυτή την έννοια μπορεί να μας δώσει την ε, εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, ε, την αυτοεκτίμηση, την ένταξη στην κοινωνία και αυτά είναι πράγματα τα οποία ε, πραγματικά δεν μπορούν να αξιολογηθούν παρά μόνο θετικά, δεν έχουν τιμή αυτά τα πράγματα. Ε, είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό να ε, προωθήσουμε τους νέους κυρίως, να τους παροτρύνουμε να ασχοληθούν με τον εθελοντισμό, κυρίως τους νέους που βρίσκονται, που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και θέλουν να εγκαταλείψουν το σχολείο. Είναι σημαντικό να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις ε, στον τομέα αυτό. Ποιοι είναι, πρέπει να παρακολουθήσουμε το φαινόμενο, ποιοι είναι οι εθελοντές στην Ευρώπη, προς τα που ε, προσανατολίζονται. Οι εθελοντές είναι οι ίδιοι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Γνωρίζουμε ότι η απάντηση είναι αρνητική. Ε, ο εθελοντισμός και η εμπλοκή με τον εθελοντισμό ε, εξαρτάται άμεσα από την κοινωνία, τις κοινωνικές και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες κτλ. Οι πραγματικότητες νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε όλο το εύρος του εθελοντισμού, δηλαδή κοινωνικών, πολιτιστικό, ψυχαγωγικό, όλα αυτά θα πρέπει να τα βοηθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ ο Σαντιάγκο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Και εγώ θέλω να προσθέσω τη φωνή μου στα συγχαρητήρια προς τον Μάρκο, διότι πιστεύω ότι πέρα από το ότι είναι ειδικό για αυτό το θέμα έκανε και εξαιρετική δουλειά. Διάβασα τα σημεία που θα ήθελα να υπογραμμίσω σε σχέση με τα όσα είπε η κυρία Ντόβα, σε σχέση με τα φορολογικά κίνητρα στι ΜΚΟ και στι εθελοντικές οργανώσεις. Αν μπορούν να επεκταθούν σε μια φορολογική αντιμετώπιση Ας το πω σε σχέση με τους ίδιους τους εθελοντές. Υπάρχουν εθελοντές που εισπράττουν πολύ μικρά ποσά και αποτελούν μέρος αυτής της λέσχης, της ομάδας. Έχω υπόψη για παράδειγμα και αθλητικές ενώσεις ή συλλόγους. Μπορεί να είναι και άλλες ενώσεις ή σύλλογοι. Τίθεται ένα πρόβλημα εδώ Πρέπει όταν αυτά τα άτομα ε, φεύγουν από αυτές τις υπηρεσίες, αυτά αυτές οι λέσχες έχουν πολύ σημαντικό πρόβλημα φορολογικό και δεν μπορούν να καλύψουν τις, ε, ε, τα ποσά πρέπει να πληρώσουν. Και έτσι πολλοί πρέπει να κλείσουν, πολλοί σύλλογοι και λέσχες ερασιτεχνών. Αναφέρομαι όχι σε σημαντικές ενώσεις και συλλόγους αθλητικές και αθλητικούς, αλλά σε εθελοντική βάση ενώσεις και συλλόγους που πληρώνουν εκεί πολύ μικρά ποσά όσοι συμμετέχουν. Να μπορεί να υπάρχει μέσα στο πλαίσιο εθελοντών ένα είδος ε, ξεχωριστού καθεστώτος για αυτά τα άτομα φορολογικά. Επίσης σίγουρα ικανοποιούμε για το ότι αυτό το θέμα έχει προωθηθεί διότι πάνε στα βουνά με τα παιδιά, κάνουν ε, καταδύσεις ε, έχουν τέτοιες δραστηριότητες αθλητικές όταν υπάρχει ένα ατύχημα μπορεί να υπάρξει μια κύρωση και πολύ σημαντικές δαπάνες ε, λόγω των προστήμων παρότι κάνουν τη δουλειά τους είναι λοιπόν θεμελιώδες να υπάρχει μια ασφάλιση, ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο που θα καλύπτει τέτοιους κινδύνους για αυτούς τους εθελοντές ευχαριστώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα συγχαρητήρια στον Μάρκο για την εξαιρετική δουλειά μια μικρή ερώτηση θα είχα για το σημείο 8 της έκθεσης. Λέει, εκπροσωπεί την άποψη ότι μέσω εθελοντικών δραστηριοτήτων οι δεξιότητες που ε, μαθαίνουν, αποκτούν ε, τα νέα άτομα θα πρέπει να εντάσσονται μέσα στο SCS. Δεν γνωρίζω τι σημαίνει αυτό. Τι ακριβώς εννοείται. Δεν εννοείται αυτό το οποίο είπατε, έτσι δεν είναι. Αυτό που ήθελα εγώ και αυτό το οποίο εγώ ζητούσα είναι οι εθελοντικές δραστηριότητες να μπορούν να πιστοποιούνται στο τέλος τέλος ότι ο Α, ο Β συμμετείχε σε αυτήν την άλλη δραστηριότητα ώστε να μπορεί να εντάσσονται, να εγγράφονται όλα αυτά σε ένα υφιστάμενο ευρωδιαβατήριο, Europass. Υπάρχουν διπλώματα πιστοποιητικά τα οποία έτσι εκδίδονται και όταν τότε το 2005 περάσαμε αυτή την ε, ρύθμιση Θέλαμε επίσης η δραστηριότητα αυτή σε μια εθελοντική δραστηριότητα να μπορεί να εντάσσεται επίσης σε αυτό το πλαίσιο παρόμοια. Δεν το έκανε τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να διευρύνουμε αυτό το εδάφιο λοιπόν, αυτή τη ρύθμιση. Αν έχουμε τελείω διαφορετική αντιμετώπιση στην επίσημη και στην ανεπίσημη ας το πούμε έτσι κατάρτιση, αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε καταλάβει τα προβλήματα. Πρέπει να διατυπωθεί και να προσαρμοστεί έτσι αυτό το άρθρο ώστε να ανταποκρίνεται στη σημερινή πραγματικότητα. Θεωρεί δηλαδή ότι μέσω των εθελοντικών δραστηριοτήτων, τα όσα αποκτούν ω δεξιότητε και ικανότητε οι νέοι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να εγγράφονται σε ένα τέτοιο διαβατήριο, ευρωδιαβατήριο. Λοιπόν, αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάποιο από την Επιτροπή θέλει να παρέμβει. Όχι. Μάρκο, εσύ έχει τον λόγο. Να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσία της βεβαίως αστειευόμενος το λέω αυτό. Λοιπόν, το σημείο 8 το οποίο υπογράμμισε και στο οποίο αναφέρθηκε η Πρόεδρος. Αναφέρεται σε αυτό το πρόβλημα της αναγνώρισης η Ευρωπαϊκή ε, ε, Επιτροπή, ε, μια και υπήρξε πρόβλημα με το Europass, έκανε πρόταση να μπει στο σύστημα πιστοποίησης. Τέλος πάντων, εμείς προσπαθήσαμε ε, να το αναφέρουμε όπως, ε, είχε, ε, το είχαμε ζητήσει από την αρχή, έστω και αν η γνώμη της Επιτροπής ήταν αρνητική. Κατά τα λοιπά, πιστεύω ότι όσα είπαν οι συνάδελφοι με ευχαριστεί, άρα να τους ευχαριστήσω για την συμβολή τους, την οποία έχουν ήδη δώσει ούτως ή άλλως από τις επισημάνσεις που έκαναν στην προηγούμενη συνεδρίαση και που προσπάθησα να τις εντάξω τις επισημάνσεις αυτές στην έκθεση και βεβαίως θα λάβει υπόψη μου και τις τροπολογίες που θα υποβληθούν ε, στις επόμενες εβδομάδες. Πάντως έχω την αίσθηση ότι συνενετικά θα προχωρήσουμε και θα έχουμε μια ενωτική στάση γιατί πιστεύω, όπως είπα και προηγουμένως, ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα που μπορούμε να στείλουμε στον κόσμο του εθελοντισμού. Ευχαριστώ λοιπόν ε, για μια ακόμα φορά τους συναδέλφους ε, για τα λόγια τους, για τα όσα έκαναν μέχρι τώρα και όσα προτίθενται να κάνουν ε, και νομίζω ότι προχωράμε καλά με αυτή την έκθεση. Εγώ θα καταθέσω μια τροπολογία για την παράγραφο 8 δεν ξέρω, μπορεί να το απορρίψει όχι η Κομισιόν. Δεν ξέρω. Αλλά δεν μπορεί να μπει μέσα στο σύστημα η CTS. Και ουσιαστικά λοιπόν είναι εσφαλμένο. Δεν είναι δυνατόν να γίνει. Μόνο αν ζητήσουμε να περιληφθεί στο ευρωδιαβατήριο. Αν δεν θέλουν, τότε να το αιτιολογήσουν η Κομισιόν. Εννοείται. 5 ενάτου είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Καλύτερα βέβαια να τα κάνουμε πριν από το καλοκαίρι για να μην τα λησμονήσουμε. Και 17, με συγχωρείτε, ναι, 17 Οκτωβρίου ψηφίζουμε. Είστε σύμφωνε και σύμφωνοι. Ωραία. Τότε προχωρώ στο επόμενο θέμα της ημερησίας τη διατάξεω. Προσβασιμότητα των ιστοτόπων οργανισμών του δημοσίου τομέα. Κύριε Μπάγκο, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω για την πολύ θετική συνεργασία που προσφέρθηκε από τους συμβούλους του ΕΛΚΑ και τα μέλη της Γραμματείας. Σίγουρο είναι ότι η πρόταση για την προσπελασιμότητα σε σχέση με αυτή την οδηγία υπευλήθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 3 Δεκεμβρίου 2012 τότε κατατέθηκε. Αυτή η οδηγία λοιπόν τι έχει υπόψη. Έχει υπόψη να μπορέσουν οι ιστοσελίδες δημόσιων οργανισμών, κρατικών οργανισμών και φορέων να είναι προσπελάσιμες για το κοινό. Να μπορούν δηλαδή ενιαίες απαιτήσει να ισχύουν όσον αφορά τις 12 ας το πω έτσι διαφορετικές δυνατότητες που προβλέπονται και αυτή η οδηγία υποστηρίζει λοιπόν την προσπελασιμότητα στα κριτήρια που ισχύουν για την προσπελασιμότητα στις ιστοσελίδες και σε σχέση ακριβώς και με τις ανάγκες ατόμων με ειδικέ ανάγκες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ατόμων με αναπηρία. Πρέπει να διασφαλίζουν τα κράτη-μέλη ότι οι ιστοσελίδες που θα συνιστώνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να είναι προσπελάσιμες για αυτούς τους ανθρώπους, διότι αυτές οι ιστοσελίδες θα βοηθήσουν αυτά τα άτομα να ζήσουν μια πιο αξιοπρεπή και καλύτερη ζωή με πιο ικανοποιητικές αναβαθμισμένε υπηρεσίες. Η προσέγγιση αυτό, αυτή στο επίπεδο των κρατών μελών δεν συντονίζεται σήμερα και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Ω εισηγητή, επιτρέψτε μου να δώσω μια περίληψη ε, εν συντομία των ε, όσων προτείνονται και σε σχέση και με τις τροπολογίες. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω με τα είδη, 12 είδη ιστοσελίδων που υφίστανται και που ε, βρίσκονται μέσα σε αυτές τις προτάσεις. Η 12η αφορά μόνο ένα συγκεκριμένο εύρος ε, τομέων, δημόσιων τομέων και επεξηγείται ότι καθιστώντας ε, προσπελάσιμες αυτές τις ε, ιστοσελίδες θα υπάρχει μια επίπτωση ντόμινο, μια ας το πω έτσι εποφελής επίπτωση και σε άλλες τέτοιες ιστοσελίδες. Να κάνω μια προσθήκη. Υπάρχει όμως μια διαφοροποίηση μεταξύ ιστοσελίδων με πολιτισμικό ή εκπαιδευτικό περιεχόμενο και αυτή τη στιγμή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτείνει εφαρμογές για τον τριτογενή τομέα, δηλαδή την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή πανεπιστήμια και σε σχέση με, τα, ε, με τις πτυχές αυτές που πρέπει να ε, λαμβάνονται υπόψη πρέπει να διαφοροποιούμαστε λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες αλλά όλων των ατόμων. Άλλα άτομα έχουν προβλήματα όρασης, άλλοι έχουν πρόβλημα ε, χρήσης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Υπάρχει ο κίνδυνος να απομονωθούν αυτά τα άτομα. Αν δεν διευκολύνουμε την προσπελασιμότητα τότε θα ζουν μια πιο απομονωμένη και πιο μοναχική ζωή Πράγμα που πρέπει να αποφύγουμε. Γι' αυτό θα πρότεινα οι αρμόδιοι φορείς να εκπονήσουν φιλικές προς τους χρήστες τεχνολογίες που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται εξίσου εύκολα και από ηλικιωμένους. Θα ήθελα να ζητήσω συνάδελφοι να υποστηριχθεί η πρόταση αυτή για, αυτό, για αυτή τη συμπλήρωση, για αυτές τις συμπληρώσεις και προσβλέπω στα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Από την άλλη τώρα πλευρά, η πρώτη ανταλλαγή απόψεων ε, ήδη ολοκληρώθηκε από πλευράς Επιτροπής ε, ΙΜΚΟ. Καταθέσαμε μια σειρά τροπολογιών από κοινού με διάφορους ε, άλλους ευρωβουλευτές συναδέλφους μας ε, μαζί με την κυρία Ναγκόμες, ε, Ρομπέρτα Αντζελίλη και άλλους. Όλα αυτά ως προσθήκες στις, στην έκθεση Χατζημαρκάκη όπως την αποκαλούμε οι τροπολογίες ε, που ε, καταθέσαμε συμπληρωματικά έχουν λοιπόν με, ε, ως εξής. Πιστεύουμε ότι η ασφάλεια και η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει όλο και μεγαλύτερη σπουδαιότητα. Θα θέλαμε στην έκθεση ΙΝΚΟ να αναφέρονται τα προβλήματα των πιο ηλικιωμένων ατόμων και όσον αφορά και την προσβασή τους σε αυτές τις υπηρεσίες. Θα θέλαμε να εξειδικευθούν περαιτέρω οι απαιτήσει ώστε να υπάρχει και να διασφαλίστε η προσπελασιμότητα αυτών των ιστοσελίδων και θα θέλαμε να εξειδικευθεί περισσότερο και το περιεχόμενο αυτών τονίζοντας την ε, σπουδαιότητα μιας ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής πολιτικής χρήσης, ε, πολιτικής χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων με την ε, ημερήσια διάταξη θεματολόγιο δηλαδή για τα ψηφιακά, την ε, ε, νεολαία ε, σε κινητικότητα, Youth in Motion και άλλες τέτοιες δράσεις. Η δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την κινητικότητα ακριβώς και τις αναπηρίες εμπεριέχει κάποια στοιχεία που θα θέλαμε να τονίσουμε, να υπογραμμίσουμε εδώ. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να αναφέρεται η νοηματική γλώσσα και αυτό μάλιστα σε αρκετά σημεία να, να συμπεριλαμβάνεται και αυτή. Με, αυτό... με αυτές τις προτάσεις θέλουμε να αναδιαμορφώσουμε, να τροποποιήσουμε το έγγραφο ώστε να συμπληρωθεί όπως χρειάζεται. Ώστε για το σχέδιο οδηγίας για την προσπελασιμότητα αυτών των ιστοσελίδων από πλευρά των κρατικών φορέων, ναι μεν τα πράγματα βαίνουν καλώς, αλλά θα πρέπει να συμπληρωθούν μελλοντικά ώστε να συμπεριλαμβάνονται όλοι οι δημόσιοι φορείς όπου και αν βρίσκονται. Σας ευχαριστώ και προσβλέπω στις παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος ΠΑΚ. Ποιος ή ποια επιθυμεί. Ευχαριστώ. Δεν έχει μικρόφωνο η κυρία ΠΑΚ, δεν τα ακούμε όλα όσα λέει. Τώρα έχει. Μέχρι τώρα κανείς δεν ζήτησε το λόγο. Άρα θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Ίσως η Κομισιόν μπορεί να τοποθετηθεί. Ορίστε, έχετε το λόγο. Ο κύριος Γένσεν Κέρστενσεν, δεν είστε εσείς. Α, λέγομαι Γιώργος Και σας ευχαριστώ που προσφέρετε την ευκαιρία στην Κομισιόν να θέσει υπόψη σας κάποιες πρώτες σκέψεις. Πρώτα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Επιτροπή σας για το επικοδομητικό έργο που έχει επιτελέσει και την σε βάθος κατανόηση του θέματος σε ό,τι αφορά ειδικότερα τον στόχο της προτάσεως σαφώς συμβαδίζουμε και σε ό,τι αφορά τις τεχνικές λεπτομέρειες, όντως έχετε καταθέσει επικοδομητικές προτάσεις, τις οποίες θα μελετήσουμε και εμείς προσεκτικά. Ευχαριστώ και την Επιτροφή σας και τον εισηγητή. Ασφαλώς και μας βρίσκουν σύμφωνους οι προσπάθειες που γίνονται η πρόταση αυτή να ενταχθεί ακόμα πιο καθαρά στην συμπερίληψη, στην πολιτική της συμπερίληψης, στην κάλυψη αναγκών ε, ανθρώπων που έχουν ειδικές ανάγκες. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι εάν όλα αυτά θα πρέπει να ενταχθούν στην συγκεκριμένη αυτή πρόταση ή αν θα πρέπει να καλυφθούν και ενδεχομένως από άλλα ξεχωριστά μέτρα. Ένα ίσονο σημασία σχόλιο έχει σχέση με το ότι το οπτικό ακουστικό περιεχόμενο, όπως λέτε και στο άρθρο 1, καλύπτεται ήδη από τις τεχνικές απαιτήσεις της προδιαγραφής ε, ΟΕΓΑΣ 0.2 και το καλύπτει και η οδηγία ίδια. Και όσον αφορά τις προτάσεις για διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής, δεν είστε το μόνο όργανο που προτείνεται να περιλάβουμε τέσσερις ακόμα τύπους ιστοσελίδων του δημοσίου τομέως, καθώς και άλλα περιεχόμενα και άλλους τύπους περιεχομένων. Η ιδέα της Κομισιόν ήταν να γίνει η πρόταση στενή αλλά αποτελεσματική, ώστε να αποφευθεί η πρόσθετη επιβάρυνση χωρών που την εφαρμόζουν. Η δε νομική βάση για την πρόταση είναι ο κατακαιρματισμός της αγοράς. Εμείς λοιπόν εξετάζουμε το τι είναι απαραίτητο για να γίνει πιο σφιχτή η αγορά που όπως εξήγησα είναι πολύ κατακαιρματισμένη και η οποία περιέχει πολλές ανασφάλειες και από την άποψη της ε, προσφοράς και της ζήτησης και εκατέρωθεν των συνόρων αλλά και στην αγορά την ίδια. Η πρόταση βασίζεται στην ιδέα ότι εάν καλύψουμε αυτούς τους 12 τύπους ιστοσελίδων που θα πρέπει κανονικά να διαθέτουν όλες οι χώρες και που προσφέρουν υπηρεσίες στους πολίτες, θα έχουμε αρκετή κρίσιμη μάζα και από εκεί και πέρα τα spillover, δηλαδή ε, οι αντίκτυποι σε άλλες ιστοσελίδες που προσφέρουν υπηρεσίες στους πολίτες θα είναι αυτόματη λίγο πολύ. Επίσης υπάρχει και ένα θέμα το οποίο ακόμα δεν έχουμε επιλύσει αλλά διαισθανόμεθα ότι ίσως υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ των τροπολογιών 6 και 10 όχι τόσο στον στόχο τους αλλά στο γεγονός ότι η μία προτείνει στις χώρες μέλη να επεκτείνουν τις διαδραστικές διαδραστικούς ιστοτόπους και στους ιστοτόπους πολιτιστικού περιεχομένου ενώ η άλλη λέει ότι η οδηγία η ίδια θα πρέπει να καλύπτει ιστοτόπους ή ιστοσελίδες με πολιτιστικό περιεχόμενο. Εδώ χρειάζεται κάποια περισσότερη μελέτη κατά τη γνώμη μας ώστε να υπάρξει μια μεγάλη επικάλυψη μεταξύ των δύο προκαλώντας τον κίνδυνο να προκύψουν αντιφάσεις. Να προτείνεται δηλαδή από τη μια μεριά το ένα πράγμα και να επιβάλλεται υποχρεωτικά από την άλλη. Πάντως, εν τέλει ευχαριστούμε για τις επικοδομητικές προτάσεις και τροπολογίες και όπως είπα θα τις μελετήσουμε προσεκτικά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, κυρία Πακ, ευχαριστώ. Εδώ φαίνεται να συμφωνούμε όλες και όλοι, άρα λύγει και αυτό το θέμα της ημερησίας διατάξεως. Όπως και πριν, 5 Σεπτεμβρίου η προθεσμία καταθέσεων τροπολογιών και 17 Δεκάτου η ψηφοφορία. Το 11 τώρα τα διάφορα. Υπάρχουν διάφορα. Όχι. Εδώ λοιπόν λίγη η κανονική συνεδρίαση. Εύχομαι σε όλες και όλους τους συναδέλφους που δεν είναι υποχρεωμένες να παραμείνουν ή και δεν τους επιτρέπεται ενδεχομένω να περάσουν καλές διακοπές. Θα τα πούμε το αργότερο στις 5 Σεπτεμβρίου για να συζητήσουμε budget amendments και budget opinions και βεβαίως τότε να έρθετε διότι μπαίνουμε πλέον σε πολύ ουσιώδη θέματα. Και σε εσά εκεί στα ορεινά σας εύχομαι επίσης καλές διακοπές όπως είπα, κλείνει τώρα η συνεδρίαση. Μόνο οι διερμηνείς επιτρέπεται να παραμείνουν και θα μιλήσουμε τώρα για το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Σύντομη συζήτηση με τους σκιώδεις εισηγητάς. Ευχαριστώ και την Κομισιόν και ωραί βουάρ. Äh, ja, ich kann nicht warten, bis die Frau kommt.